σημαντικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να εξυπηρετηθούν οι στόχοι των Ηνωμένων Εθνών ώστε να μπορέσει η κατάσταση αυτών των ανθρώπων να βελτιωθεί. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τον ε, κύριο Συγητή, τον συνάδελφο κύριο Σαλαφράγκα. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, μου είναι χειρίστη μία πρόταση ψηφίσματο για την περάτωση αυτή τη συζήτηση. Η κοινή συζήτηση έληξε. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στι 12 το μεσημέρι. Το επόμενο σημείο στη μερίσια διάταξη είναι δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής με θέμα θύματα πυρκαγιών που σημειώθηκαν πρόσφατα σε υφαντουργία, ειδικότερα στο Μπανκαλαντές. Η ε, Υπουργό, η κυρία ε, Λουσίντα Κρέιτον, έχει το λόγο εξ του Συμβουλίου. Minister, the floor is yours. <laughs> mr um, president uh, honourable members αγαπητά μέλη οι πρόσφατες πυρκαγιές ε, κοντά στη Ντάκα, στην Ασούλια, αποτέλεσαν μια μεγάλη τραγωδία. Ε, περισσότερο από 100 άτομα βρήκαν το θάνατο σε αυτή την ε, τεράστια πυρκαγιά και όλοι εκφράσαμε τη, τον αποτροπιασμό μας για όλους αυτούς που έχασαν ε, άτομα της οικογένειας. Αυτό το συμβάν δείχνει ένα ευρύτερο πρόβλημα που υπάρχει σε πολλά εργοστάσια στο Μπαγκλαντές γιατί δεν υπάρχουν βασικοί κανόνες ασφαλείας. Δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτό το συμβάν ασχολίαστο. Θα πρέπει να ζητήσουμε από τις αρχές ε, του Μπαγκλαντές να προωθήσουν αρχές ασφαλείας και εποπτείας. Όλοι όσοι εργάζονται στα εργοστάσια ηματισμού έχουν βασικά δικαιώματα για να εργάζονται εν ασφαλεία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο γιατί είμαστε ο σημαντικότερος εταίρος του Μπαγκλαντές και βεβαίως θα πρέπει να δημιουργηθούν ναι, πολλές θέσεις εργασίας. Ο τομέας της ένδυσης είναι πολύ σημαντικός για το Μπαγκλαντές, για τις εξαγωγές τους μέσα στα πλαίσια της αγοράς χωρίς ποσοστώσεις και χωρίς δασμούς που, προσφέρει, που προσφέρεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στα πλαίσια του γενικού καθεστώτος δασμολογικών προτιμήσεων. Αλλά τη στιγμή που παράγονται αγαθά σε εργοστάσια με πολύ χαμηλές προδιαγραφές ασφαλείας και τη στιγμή που διατρέχουν κίνδυνο οι εργαζόμενοι στην καθημερινή τους εργασία, θα πρέπει να αντιδράσουμε. Γι' αυτό ζητάμε βελτιώσεις στις προδιαγραφές εργασίας, στο χώρο εργασίας. Θέλουμε οι εργοδότες να μπορέσουν να ανταποκριθούν στους κανόνες υγείας και ασφάλειας και το έχουμε δει και με εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου. Αλλά η τραγική πυρκαγιά ε, κατέδειξε ότι θα πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μία ε, σειρά μηχανισμών για να αντιμετωπίζονται αυτά τα ζήτηματα, όχι μόνο στο Μπαγκλαντές. Θα ήθελα να εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτούς τους μηχανισμούς σε σχέση με τις αρχές του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Το ε, σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων είναι ένα από τα βασικά μας μέσα για να συνδέσουμε τα κοινωνικά ζητήματα με τα ε, ζητήματα που άπτονται της ασφαλείας και με, μέσα στα πλαίσια του GSP+. Δηλαδή μιλάμε για προτιμησιακές εμπορικές σχέσεις με βάση 27 διεθνείς συμβάσεις που περιλαμβάνουν και δικαιώματα στην εργασία και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Όλες αυτές οι προτιμησιακές συμφωνίες μπορούν να αποσυρθούν σε χώρες όπου υπάρχει ε, διακύβευση και μη τήρηση των συμβάσεων. Δεν πρόκειται για κενό γράμμα. Συνέβη σε πολλές περιπτώσεις όπως τη Λευκορωσία και το Μιανμάρ όταν αποσύρθηκαν, ε, ε, αποσύρθηκε το GSP+. Και αυτό έγινε και στη Σρι Λάνκα. Μας ενδιαφέρει η προώθηση των περιβαλλοντικών προδιαγραφών και για να φτάσουμε σε αυτούς, στην τήρηση αυτών των μέτρων θα πρέπει να προωθήσουμε όχι μόνο διμερείς αλλά και πολυμερείς σχέσεις μέσα στα πλαίσια του ΠΟΕ. Έτσι, στις διμερείς εμπορικές σχέσεις προωθούμε και προδιαγραφές βιωσιμότητας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν δραστηριοποιούμαστε και ευρύτερα. Μας ενδιαφέρει να ανταποκριθούμε στις προδιαγραφές του ΠΟΕ και του ΔΟΕ και γνωρίζουμε ότι υπάρχει και περιβαλλοντικό και κοινωνικό ντάμπινγκ γιατί υπάρχει στρέβλωση των κανόνων ανταγωνισμού. Χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα που είναι διαθέσιμα καθώς και τις ε, ρήτρε ε, βιώσιμης ανάπτυξης έτσι ώστε να αναχαιτήσουμε αυτούς τους κινδύνους. Μια άλλη βασική πτυχή ε, είναι οι επενδύσεις οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που επενδύουν στο Μπαγκλαντές δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Μπορούν να βελτιώσουν και τις συνθήκες εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι ε, φέρουν συγκεκριμένη εταιρική ευθύνη κατά την απασχόληση σε τρίτες χώρες. Η εταιρική σχέση και ευθύνη είναι ύψης της σημασίας και θα ε, ανταποκριθούμε και στην τελευταία ανακοίνωση της Επιτροπής. Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, η πυρκαγιά στον Μπαγκλαντές θα πρέπει να αποτελέσει προειδοποίηση για μας. Δεν μπορούμε να ε, θέτουμε σε κίνδυνο τις ζωές των εργαζομένων. Θα πρέπει να προωθήσουμε τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας και να χρησιμοποιήσουμε το GSP τις ε, προτιμησιακές σχέσεις έτσι ώστε να τηρούνται οι σωστές προδιαγραφές. Θα πρέπει να συνεργαστούμε και μέσω του ΠΟΕ και του ΔΟΕ για να ε, εφαρμόσουμε τις αρχές ασφάλειας και οι επιχειρήσεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να αποτελούν μια θετική δύναμη για να επιβάλλουν τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφαλείας σε αυτές τις χώρες. Θα εργαστούμε ε, στενά έτσι ώστε να αποτραπούν τέτοιες, τέτοια συμβάντα όπως η πρόσφατη πυρκαγιά στο Μπαγκλαντέ. Ευχαριστώ την εκπρόσωπο της, ε, εκπροσώπου για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Now I'll give the floor to Commissioner. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Επίτροπο Κρυσταλίνα Γεωργίευα, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές. Κύριε Υπουργέ Κρέιτον, όπως ακούσαμε και από την Υπουργό, η πυρκαγιά στο Ευθυντεχνείο Ενδυμάτων ε, στην Αστούλια, στο Μπαγκλαντές, έβαλε στο επίκεντρο ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει σε πολλά άλλα μέρη. Το πρόβλημα δηλαδή των ελλείψεων και των αδυναμιών σε ό,τι αφορά την οθέτηση και την εφαρμογή κοινωνικών προτύπων και κανόνων, ιδίω ε, στην ε, Νότια Ασία στον τομέα των ειδών ένδυση. Και σίγουρα πρέπει να αποτίσουμε φόρο τιμή στα θύματα, όχι μόνο εκείνο το τραγουδιών, αλλά και πολλών άλλων. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο αν θέσουμε σε Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το ζήτημα ε, στις σχέσεις μας με τους μα μας και αν αναλάβουμε συγκεκριμένη δράση. Ακριβώς αυτό είμαστε αποφασισμένοι να πράξουμε και το πράττουμε ήδη. Θα ήθελα να, φέρω, να, να θέσω υπόψη σας συγγνώμη τι έχει γίνει έκτοτε. Πρώτον, στην ΤΑΚΑ οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έδρασαν τάχιστα. Την επόμενη μέρα τη πυρκαγιά, ένα σχέδιο το οποίο συγχρηματοδοτείται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Γερμανία για την βελτίωση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών κανόνων στα εργοστάσια, για την παροχή ατροφαρμακευτική περίθαψη ε, και τροφίμων ε, και άλλων στου πληγέντε, τέτοια σε ισχύ. Και επίση ε, υπήρξε και κοινό, και κοινό λυπητηρίων από όλου του πρέσβει, όπου έδειχνε ότι μας, μας ενδιαφέρουν όλα τα κοινωνικά ζητήματα και ιδίως το θέμα της ασφάλειας στα θέματα που αφορούν τις επάπτωτες των εμπορικών σχέσεων. Πρέπει να πούμε ότι το Μπαγκλαντές ε, έχει ως βασικό κύριο εμπορικό εταίρο την Ευρωπαϊκή Ένωση, 57% των ε, εξαγωγών έρχονται στην Ένωση και κυρίως πρόκειται για είδη ένδυσης. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό για, τους, για τις επιχειρήσεις μας, για τους καταναλωτές μας και την κοινωνία μας. Όλα αυτά που συμβαίνουν στο κοινωνικό επίπεδο στον Παγκλαντές. Δεύτερον, συνεχώς βάζουμε τα μεγκληματική υγεία, την ασφάλεια στο επίκεντρο. Παραδείγματο χάρη έχουμε την, ε, το πρόγραμμα για αξιοπρεπή εργασία του Διεθνούς γραφείο Και έχουμε στηρίξει ε, την δημιουργία σχετικών προγραμμάτων και στον Μπαγκλαντές Όπω παραδείγματο χάρη βοήθεια σε αρχέ, τη ενό εργοδοτών για να γίνονται έλεγχοι συμμόρφωση ε, στα εργοστάσια. Και θέλουμε να βοηθήσουμε επίση και στην εκπαίδευση των επιθεωρητών εργασία. Εργαζόμαστε επίσης ε, και με την Διεύθυνση Αστικής Πολιτικής Προστασίας και Υπηρεσιών της πυροσβεστική των Μπαγκλαντές. Τρίτον, ο πρέσβης μας, ε, William Hanna, συναντήθηκε με εκπροσώπους ε, της ε, Ένωσης των παραγωγών και εξαγωγών ειδών ένδυση στο Παγκλαντές για να συζητήσει τη συνεργασία τους σε θέματα ασφάλειας των εργοστασιών στον τομέα του Πρεταπορτέ. Και επίσης η συζητάμε τα θέματα της ε, ασφάλειας, θα τα δούμε και στις αρχές του 2013 που θα έχουμε μια συζήτηση σε επίπεδο των αρχηγών αντιπροσωπιών της Ένωσης για το θέμα της ένδυσης. Επίσης δεσμευόμαστε για να προωθήσουμε και να υλοποιήσουμε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα κοινωνικής ευθύνης. Τα είπε και η Υπουργός. Θέλουμε λοιπόν κάποιες γενικές κατευθύνσεις ε, να υιοθετήσουμε και στο διάλογό μας με τις ε, αρχές του Μπαγκλαντές. Αυτό ήδη έχει συμβεί και στην ε, συνεδρία της Κοινής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Παγκλαντές το Δεκέμβριο συγκεκριμένα. Όχι μόνο τότε όμω, αλλά είναι συστηματικά ένα θέμα το οποίο αναφέρουμε σε επαφέ μα με τι αρχέ του Μπαγκλαντέ, δηλαδή βελτίωση των συνθηκών εργασία. Είναι ένα θέμα που το αναφέρουμε συνέχεια, όπω το 2011. Οπότε και διοργανώσαμε στην ΤΑΚΑ ένα σεμινάριο για την αξιοπρεπή εργασία. Εκεί υπήρξαν εκπρόσωποι όλων των κλάδων και διαβιβάστηκαν στην κυβέρνηση του Μπαγκλαντέ οι συστάσει, οι οποίε δείχνουν και τι ανησυχίε που εκφράζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπω παραδείγματο χάρη ε, στο ψήφισμα της 8 Ιουνίου του 2011 για την εξωτερική διάσταση της κοινωνικής πολιτικής. Κάτι πιο γενικό είναι ότι Ευρωπαϊκή, ε, μάλλον το ψήφισμα της 23 Οκτωβρίου του 2012 για το μέλλον της αναπτυξής πολιτικής της Ένωσης. Εκεί ετέθη επίσης το ζήτημα της ανάγκης να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές ανισότητες εν ώψη της ε, αύξησης της οικονομίας πρέπει να επωφεληθούν και τα φτωχότερα στρώματα από την άνθηση του τομέα της ένδυσης ε, στη χώρα. Αυτό θα βοηθήσει και αυτό το έχουμε συμπεριλάβει στον ε, ε, ολοκληρωμένο διάλογο που έχουμε με τον Μπαγκλαντές. Θα ήθελα λοιπόν να, να συνοψίσω λέγοντας ότι πρόκειται για μια υπόθεση η οποία προσέλκυσε τη διεθνή προσοχή και σίγουρα προσέλκυσε την έντονη προσοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί έχουμε ειδικές σχέσεις με το Μπαγκλαντές αλλά και ε, με άλλες χώρες. Το Πακιστάν για παράδειγμα και εκεί ε, ξέσπασε μια πυρκαγιά, παρόμοια πυρκαγιά. Ευτυχώς όμως με όχι τόσο πολλές απώλειες ανθρώπινης ζωής. Θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το γεγονό ότι παραμένετε εστιασμένοι, δείχνετε τον ενδιαφέρον σα για το θέμα αυτό και μα παρακινείτε να κάνουμε κι εμεί πάνω το δυνατόν, διότι αυτό που ε, διακυβεύεται είναι η ασφάλεια των ε, ανθρώπων στι χώρε αυτέ, αλλά όπω είπε η Υπουργό, πρέπει κι εμεί να δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ε, δύναμη του καλού και έτσι πρέπει να δράσουμε. Και αν μου επιτρέπετε, θέλω να ζητήσω συγγνώμη γιατί πρέπει να φύγω, αλλά θα μείνει ο Επίτροπο Μπαρνιέ. Θα με αντικαταστήσει επάξια. Δύο στην τιμή του ενό. κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, ανοίγει ο κύκλο των ομιλητών εξ ονόματο των πολιτικών ομάδων. Ε, είχε, für die ah για το ΕΛΚ θα λάβει τον λόγο ο συνάδελφος Τόμας Μπαν. Για τρία λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και για τα γερμανικά σας. 112 άνθρωποι αποβίωσαν κατά τη μεγάλη αυτή πυρκαγιά στην βιομηχανία αυτή ε, το 2012 και πραγματικά συγκλονίστηκαν παγκόσμια οι άνθρωποι από αυτό. Το Δεκέμβριο σχεδόν 300 άτομα θα ήταν θύματα, ήταν θύματα μιας ε, εκρήξης ε, στο Καράτσι, στο Πακιστάν. Θα μπορούσαν να ζουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι αν υπήρχαν ασφαλείς εγκαταστάσεις ε, και οι διατάξεις των, εντολέων από την Ευρώπη είχαν γίνει σεβαστές. Πολλές φορές όμως οι έλεγχοι είναι προσχηματικοί και πολύ χαλαροί. Οι υπεύθυνοι δεν τιμωρούνται, δεν προσάγονται στα δικαστήρια. Οι ευθύνε είναι μπαλάκι που μετατίθεται διαρκώς στο γήπεδο από τη μία στην άλλη πλευρά. Οι ιδιοκτήτες εργοστασίων και επιχειρηματίες είναι εκείνοι οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται και εκείνοι που έχουν ε, τις ε, αγοράζουν αυτά τα προϊόντα στην Ευρώπη ε, έχουν ιδιαίτερα ευνοϊκές τιμές για τα εμπορεύματα που αγοράζουν. Θα έπρεπε να μπορούν να είναι ασφαλείς οι θέσεις απασχόλησης εκεί. Πολλά έκανε τον Μπαγκλαντές μέχρι σήμερα, ιδιαίτερα για την καταπολέμηση της εργασίας των παιδιών στον τομέα της κλωστοϊφαντουργίας για παράδειγμα. Πρέπει να τα αναγνωρίσουμε αυτά. Η διατάξη διαγραφέ του Παγκοσμίου του Διεθνού Γραφείου Εργασία πρέπει να τηρούνται όμω και να είναι σεβαστέ. Οι διακηρύξει και τα λόγια δεν επαρκούν. Και τα όσα γίνονται και πρέπει να γίνουν από πλευρά τη Ευρώπη ε, μέσω των ε, όρων εργασία εκεί που πολλέ φορέ είναι ελεηνοί και για την αξία κιόλα και των περιβαλλοντικών προδιαγραφών και των κοινωνικών προδιαγραφών. Πρέπει να ασκηθεί η πίεση των καταναλωτών ως αποτελεσματικό όπλο ώστε να υπάρξουν αηφόρα αλλαγές ε, προς το καλύτερο. Όμως υπάρχουν κάποιες ε, τροπολογίες και αιτήματα υπερβολικά όπου ε, νομικές ε, παρεμβάσεις ζητούνται στο διεθνές επίπεδο. Διατάξεις διημερείς συμφωνίες και διατάξεις συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων κρατών επαρκούν. Πρέπει όμως με συνέπεια να εφαρμόζονται και να υλοποιούνται. Κυρώσει, ε, για παράδειγμα π.χ. σε σχέση με πολυεθνικές ε, εταιρείε που δεν ε, προσαρμόζονται προς αυτές τις διατάξεις. Οι καταστροφές αυτές δείχνουν ότι σε κάποιες επιχειρήσεις δεν είναι σεβαστή η κοινωνική ευθύνη. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη, εταιρική κοινωνική ευθύνη και πρέπει να είναι σεβαστή. Επιτόπου θα έπρεπε να πούμε ότι δεν αλλάζει τίποτα δυστυχώς ε, υπέρ των εργαζομένων. Ε, η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθένης είναι όμως υποδειγματική. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις συγκεκριμένα συνεισφέρουν και επομίζονται την κοινωνική τους ευθύνη. Ο εθελοντικός χαρακτήρας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης πρέπει να παραμείνει όμως. Ενθαρρύνει για ενδυναμωμένες προσπάθειες. Υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτές τις, αυτά τα μέτρα που μπορούν να συνεισφέρουν και να μεριμνήσουν για θετικές αλλαγές. Ευχαριστώ. Επόμενος αγορητής θα είναι ο συνάρφος κύριος Μπέρντ Λάγκε εξ ονόματος των Σοσιαλδημοκρατών για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, εμεί όλοι μα αγοράζουμε και φοράμε ρούχα τη εταιρεία CA, τη HM, τη Μπενετών και άλλων εταιριών που είναι μεγάλε επιχειρήσει και λαμβάνουμε πολύ λίγο υπόψη, πιστεύω, ποια είναι η αλυσίδα που οδηγεί σε αυτά τα προϊόντα. Πώς είναι δυνατόν με παιδική εργασία να, να παράγεται μαλλί και με απάνθρωπες συνθήκες ε, στο Πακιστάν, στο Μπαγκλαντές να παράγονται ενδύματα και σε υψηλές τιμές να μεταπολούνται μετά και να διατίθενται στην Ευρώπη και να μεγιστοποιείται το κέρδος αυτών των επιχειρήσεων πάντα. Εγώ πιστεύω ότι εμείς από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πρέπει να απαιτήσουμε την κοινωνική τους ευθύνη να την επομιστούν με συνεπή τρόπο και μάλιστα από πλευράς των δράσεών τους να αποδεικνύουν πώς η αλυσίδα παραγωγής ανταποκρίνεται στις διεθνείς διατάξεις και προδιαγραφές του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Και γι' αυτό ζητώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβάλλει την υποχρέωση σύνταξης εκθέσεων από πλευράς των μεγάλων επιχειρήσεων για το πώς ανταποκρίνονται στην εταιρική κοινωνική ευθύνη. Κατά δεύτερο λόγο αυτές οι επιχειρήσεις πρέπει από κοινού να δράσουν Φυσικά όταν υπάρχει ανταγωνισμός ε, και υπάρχει dumping ε, τότε μπορεί να κάνει κάθε επιχείρηση ό,τι επιθυμεί κατά το δοκούν. Εμείς πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες οι ευρωπαϊκές ε, επιχειρήσεις να υποχρεωθούν από κοινού να τηρούν αυτές τις κοινωνικές διατάξεις και προδιαγραφές. Και ζητώ να ενεργοποιηθούμε ώστε να προσαρμοστούν αυτές προς αυτές τις απαιτήσεις. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ κύριε Λάγκε. Στη συνέχεια ο συνάδελφος Μπένιον εξ ονόματος της Άλντε. Δύο λεπτά παρακαλώ. Um, yeah, thank you. Uh, Ευχαριστώ. Ζήτησα πρόταση ψηφίσματος ε, και για την πυρκαγιά στην Τάκα αλλά και στο Καράτσι να ενταχθεί δηλαδή στην ημερήσια διάταξη και χαίρομαι. Αυτό το είχα ζητήσει το Νοέμβριο. Πολλοί θα μπορούσαν να έχουν σωθεί αν υπήρχαν προδιαγραφές πυρασφάλειας. Χαίρομαι για τις προσπάθειες που καταβάλλονται για τη βελτίωση των συνθήκων ασφαλείας. Χτες ε, ε μία απόφαση μεταξύ εργαζομένων εργοδοτών και κυβέρνησης και θα ήθελα και η κυβέρνηση του Πακιστάν να αναλάβει μια παρόμοια δράση. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε τέτοιες, τέτοια ατυχήματα τη στιγμή που κλειδώνονται οι, πρώτες και, πόρτες και δεν υπάρχουν ε, οδοί διαφυγής. Πολλά θα πρέπει να γίνουν για να καταπολεμηθεί η ενδυμική διαφθορά που υπάρχει στο σύστημα επιθεώρησης. Και αυτό αφορά και τις, τη μεγάλη ευθύνη που φέρουν οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι μεγάλες μάρκες. Γιατί βλέπουμε ότι δεν ανταποκρίνονται. Δεν θα πρέπει όμως να θεωρήσουμε τις ε, πολυεθνικές ε, ηματισμού ε, ως οργανισμούς, ως φορείς που φέρουν συγκεκριμένη ευθύνη και πολλοί προσπάθησαν να αποδώσουν ευθύνη μόνο στις πολυεθνικές. Όμως η βασική ένοχη είναι οι ιδιοκτήτες βιομηχανιών και χώρων όπου ε, κατασκευάζονται τα ενδύματα αυτά. Εξ ονόματος των φιλελευθέρων και δημοκρατών θα ήθελα να τονίσω ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε τις συνθήκες ασφάλειας και υγείας και ε, θα πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση στο Μπαγκλαντές όπως ορίζει και η Κομισιόν. Με την συνάδελφο κυρία Λάμπερτ, εξ ονόματος της ομάδας των Πρασίνων, για δυόμιση λεπτά. Thank you, Chair. Σε ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ ομιλώ υπό την ιδιότητά μου ως επικεφαλής αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καλύπτει και το Μπαγκλαντές μεταξύ άλλων χωρών ως αντιπροσωπεία. Και όπως και άλλοι θέλουμε και εμείς να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας ε, προς τους οικείους ε, και συγγενείς ε, των όσων έπεσαν θύματα αυτών των πυρκαγιών σε αυτές τις βιομηχανίες κλωστοϊφαντουργίας και αλλού. Και πέρα από το Μπαγκλαντές, ενώ επικεντρωνόμαστε σε αυτό, υπάρχει αυτό το ζήτημα, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα περιθώρια κέρδους που οδηγούν σε συμπίεση όχι μόνο μπορούν να οδηγήσουν σε αυτές τις καταστάσεις αλλά και σε ε, λήψεις και ελλείμματα όσον αφορά την ασφάλεια και ανησυχούμε γιατί πολλές από τις μεγάλες ε, επιχειρήσεις που έχουν τέτοιου είδους συμβάσεις ε, δεν ήθελαν να το αναγνωρίσουν αυτό το γεγονός για παράδειγμα κατά την περίοδο όπου συνέβη αυτή η τραγωδία έχοντας κιόλας αξιολογηθεί από τέτοιου είδους ε, ελεγκτές ε, τα κτίρια αυτών των επιχειρήσεων και σε σχέση με το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές όσον αφορά τις αποζημιώσεις ε, και την περίθαλψη των οικείων όσον αφορά τα θύματα που σημειώθηκαν. Καλωσορίζουμε επίσης και τις συνεισφορές από υπερπόντιες τέτοιες εταιρείες. θα ελπίζαμε να ήταν περισσότερες αυτές οι δράσεις. Και σε σχέση με τις ε, επαφές όσον αφορά τις, ε, το Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Ε, όλα αυτά είναι θετικά για την δέσμευση να υπάρξει δραστηριοποίηση όσον αφορά τους υφιστάμενους νόμους διατάξεις ώστε να μπορέσουν να εφαρμοστούν αυτές οι διατάξεις και οι νόμοι και θα υπάρξουν επιπτώσεις αν δεν συμμορφωθούν και δεν σεβαστούν αυτές τις διατάξεις οι αρμόδιοι. Αυτό είναι καθαρά κυβερνητική ευθύνη, ευθύνη των αρμοδίων. Επίσης πρέπει να διασφαλιστεί θα υπάρχουν και ενεργά συνδικάτα και τα δικαιώματα και οι υπέρμαχοι των ε, δικαιωμάτων, των εργασιακών δικαιωμάτων ε, θα προστατεύονται. Είχαμε πρόσφατα δολοφονίες τέτοιων ε, ατόμων και θα πρέπει πραγματικά ενεργά να μπορούν να δραστηριοποιούνται τα συνδικάτα επί τόπου σε συνεργασία με, τις, με επιτροπές ε, για την ε, υγεία και την περίθαψη και την ασφάλεια πάντα να υπάρχουν και πληροφορίες για όσους δεν συμμορφώνονται με αυτές τις διατάξεις. Υπάρχει εδώ κέριος ρόλος στην βελτίωση των διατάξεων όρων και προϋποθέσεων. Εκφράζουμε την θλίψη μας ε, γιατί κάποιες επιχειρήσεις δεν ήταν καθόλου πρόθυμες να συνεισφέρουν και δεν δραστηριοποιήθηκαν όπως θα έπρεπε. Ως καταναλωτές θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι τα ρούχα τα οποία φοράμε δεν δεν έχουν ε, οδηγήσει στο να καταπατηθούν τα δικαιώματα εκείνων που παρήγαγαν αυτά τα ρούχα. Και θα πρέπει σε σχέση με το Μπαγκλαντέ και άλλες χώρες να συνεισφέρουμε ώστε να βελτιωθούν οι εργασιακέ προδιαγραφές, οι όροι και προποθέσει υπό του οποίου εργάζονται τα άτομα αυτά εκεί. Ευχαριστώ. Ε, και το λόγο τώρα έχει η κυρία Μουσκαρντίνη εξ των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών. Η τραγωδία αυτή του Μπαγκλαντές δεν είναι μοναδική. Είναι μία από, τις μεγάλες, από τα μεγάλα αυτά συμβάντα σε μία σειρά πυρκαγιών για τα οποία φέρουν ευθύνη οι αρμόδιες αρχές και οι υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων αυτών. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτανθεί στις δικές μας επιχειρήσεις που ε, έχουν εγκατασταθεί στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες έτσι ώστε να ελέγξουν τις εγκαταστάσεις στα εργοστάσια ηματισμού. Να δουν δηλαδή κατά πόσο ε, τηρούνται οι προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που εργάζονται σε αυτά τα μέρη του κόσμου με χαμηλό εργατικό κόστος θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι η παγκοσμιοποίηση και η ελεύθερη αγορά δεν μπορούν να οδηγήσουν σε σύγχυση όπου θα πλήττονται μόνο οι ασθενείς και οι φτωχοί. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο συνάδελφος κύριος Νικόλαος Σαλαβράκος εξ ονόματος της Ευρώπης Ελευθερίας και Δημοκρατίας για 1,5 λεπτό. Οι άσκοποι θάνατοι 400 περίπου ανθρώπων στις δύο πρόσφατες πυρκαγιές στα ασιατικά εργοστάσια και ιδιαίτερα η πρόσφατη πυρκαγιά στο εργοστάσιο Ταζίν στον Μπαγκλαντές πιστεύω ότι θα πρέπει να προβληματίσουν όλους τους καταναλωτές και να αποτελέσουν έναυσμα για την άσκηση πίεσης στις χώρες αυτές ως προς τις συνθήκες ασφαλείας αλλά συνάμα και για την αποκατάσταση των όρων του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Δυστυχώς, οι αυξανόμενες καταναλωτικές ανάγκες της Δύσης και ο σκληρός ανταγωνισμός αναγκάζουν τις μεγάλες εταιρείες να μεταφέρουν την παραγωγή τους σε ασιατικές χώρες, που είναι ασυναγώνιστες σε σχέση με την Ευρώπη, καθώς το μηνιαίο εισόδημα των εργατών αυτών στις περιοχές είναι 37 δολάρια. Δηλαδή κάτω από ένα ευρώ την ημέρα κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι. Με τον τρόπο αυτό απαθής εξολοθρεύουμε τις αντίστοιχες κλαδικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι αντί να αναζητούμε ανταγωνιστικούς παραδείσους εκτός Ευρώπης πρέπει να τις δημιουργούμε μέσα στην Ευρώπη και πρέπει να απαιτήσουμε να ληφθεί σε παγκόσμιο επίπεδο το ελάχιστο όριο εργατικού κόστους να είναι ανάλογο προς τις συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης οποιοδήποτε εργαζομένου. Δεν μπορεί να αφήνουμε ασίδωτες τις αγορές και να ερχόμαστε και να δινόμαστε, να ενδιόμαστε εμείς οι Ευρωπαίοι πολίτες με ενδύματα τα οποία είναι προϊόντα εκμετάλλευσης νέων ανθρώπων παιδιών τις περισσότερες φορές και πολλές φορές βαμμένα με αίμα. πρέπει να το λάβουν υπόψη τους αυτό οι έλληνες καταναλωτές αλλά πρέπει και η κομισιόν να δει πώς φορολογικά θα αντιμετωπίσουμε το θέμα με δασμούς σε αυτά τα προϊόντα. ευχαριστώ. Κύριε Εξ ονόματος ομάδας Γκουε, το λόγο έχει ο συνάδελφος κύριος Μέρφυ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχά θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στι οικογένειε των 112 εργατών που έχασαν αχρίαστα τη ζωή του ε, στο ΤΑΖΡΙΝ, το εργοστάσιο τη τεχνία ενδυμάτων ε, τον προηγούμενο Νοέμβριο, αλλά και στι οικογένειε των 700 περίπου εργατών ε, σε άλλα τέτοια εργοστάσια. Στο Παγκλαντές σε πυρκαγιές έχουν χάσει τη ζωή του από το 2006 και μέχρι τώρα. Βλέπουμε ότι η τριμερή του μπαγκλαντέ έχει βγάλει μια διακήρυξη για την ασφάλεια. Υπήρχαν όμως ήδη νομοθετήματα από το 1991, από το 2006 για την προστασία τη ευημερία, της ε, προστασία των εργαζομένων, τα οποία όμως ε, τα είχαν παραγνωρίσει και ξέρουμε ότι είναι η χώρα αυτή δεύτερη στην, ε, στις εξαγωγή ενδυμάτων. Πάρα πολύ μεγάλο ο τζίρος η Tommy Hilfiger, η ο Calvin Klein, το H&M και η Walmart ε, φτιάχνουν εκεί τα ενδύματά τους. Το 85% όμως των ε, ε, εργατών εκεί που είναι γυναίκες περισσότερες παίρνουν πάρα πολύ λίγα χρήματα το μήνα και φυσικά ελάχιστη είναι η συνδικαλισμένη κυβέρνηση του Μπαγκλαντές πολλές φορές με, ένοπλες, με, με ένοπλους διασπά και διαλύτης διαδηλώσεις τους. Και πολλές φορές ε, ε, υπάρχουν και βουλευτές οι οποίοι έχουν, ε, είναι ιδιοκτήτες εργοστασίων δημάτων. Αυτοί λοιπόν θα πρέπει να είναι και οι ένοχοι, όσοι είναι οι ιδιοκτήτες αυτών των παγίδων θανάτου που αποτελούν αυτά τα εργοστάσια είναι ανήθικοι, ε, δεν τηρούν κανένα, ε, κανένα κώδικα διοντολογία, αλλά και όχι μόνο οι όλες οι πρακτικές που γίνονται στο Μπαγκλαντές, στο Πακιστάν, ε, ενέχουν σημαντικούς κινδύνους, ειδικότερα ε, σε ό,τι αφορά την αμοβολή ε, που γίνεται για τα τζιν. Είναι μια πρακτική που έχει αποτέλεσμα 100 εκατομμύρια τζιν που έχουν ε, υποστεί τη διαδικασία της αμοβολής να εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε ότι αυτό όμως μπορεί να δημιουργήσει καρκίνο στους πνεύμονες, στους εργαζόμενους εκεί σε αυτά τα εργοστάσια. Πρέπει λοιπόν να το απαγορεύσουμε αυτή την πρακτική και να απαγορεύσουμε και αυτά τα τζιν. Στους άλλους εγγεγραμμένους ομιλητές, I call colleague ο κύριος Μίτσελ έχει το λόγο για τρία λεπτά. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Πρόκειται για μία ε, καταστροφική κατάσταση και τη στιγμή που μιλάμε για θέματα ε, ανάπτυξης στα πλαίσια της ΑΚΕ μας ε, αποτροπιάζει το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους κάτω από αυτές τις συνθήκες. Αλλά πολλοί λένε ότι ε, και εκφράζουν τον αποτροπιασμό τους συνεχώς και καταδικάζουν κάποιον άλλο, ιδιαίτερα τις μεγάλες επιχειρήσεις. Ε, δεν μπορούμε να πούμε ότι όλες οι επιχειρήσεις δεν τηρούν κανόνες δεοντολογίας. Αν λάβουμε υπόψη το 0,7% του δικού, του δικού μας ΑΕΠ και τους φόρους, ε, και τους φόρους που πρέπει να ε, αυξήσουμε για να φτάσουμε σε αυτό το 0,7% του ΑΕΠ, βλέπουμε ότι αυτό ισχύει προτερικά σε εμά. Δηλαδή όλοι προτρέπουν όλους να μην καταβάλουν Ε, ο τομέας του ηματισμού απασχολεί 15,3 δις ανθρώπους. Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι αν δεν τους βοηθήσουμε. Τώρα μιλάμε για ε, συγκεκριμένους προϋπολογισμούς, για ανθρωπιστική βοήθεια ε, και σφετεριζόμαστε αυτά που δεν θα έπρεπε. Νομίζω ότι τη στιγμή που μιλάμε για random auditing of the standards in these workplaces, no provide uh, ε, τη στιγμή που μιλάμε για ένα μέσο ανάπτυξης και μέσα στα πλαίσια αυτής της ε, πυρκαγιάς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από τότε που έγινε η πυρκαγιά στα Tazrin ε, Fashions έκτοτε είχαμε πληθώρα πυρκαγιών αλλού. Γι' αυτό θα πρέπει να προωθήσουμε συγκεκριμένες προδιαγραφές έτσι ώστε να μην ε, συνεχίσουμε αυτή μας την ε, πορεία. Θέλετε να απαντήσετε σε μία ερώτηση του κυρίου Μέρφη μέσα στα πλαίσια μπλε κάρτας. Κύριε Μέρφη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Υποθέτω ότι εμένα στόχευε ο κύριος ε, Μίτσελ. Γιατί θίγει πολιτικά ζητήματα και γιατί μιλάει για φόρους ε, ιδιοκτησίας και τι νόημα έχουν όλα αυτά τη στιγμή που ε, καταβάλλονται δασμοί μέσα στα πλαίσια της κυβέρνησης που υποστηρίζετε εσείς και εάν υπήρχε μία νέα φορολογική πολιτική θα σας ε, υποστηρίζαμε. Αν γινόταν κάτι τέτοιο, τότε δεν θα μπορούσε η Ιρλανδική κυβέρνηση να πληρώσει τους δημόσιους υπαλλήλους της. Θέλετε άμβλωση, έχετε την αύριο. Μην ξεχνάτε ότι όλοι ζητάν τα πάντα. Εμείς προσπαθούμε να μπορέσουμε να επιβάλλουμε τέλη και δασμούς έτσι ώστε να μην αποδίνουμε ευθύνη σε άλλους. Γιατί δεν ερχόσαστε στην Επιτροπή ΝΤΕΒΕ, ποτέ δεν σας είδα και δεν νομίζω ότι σας έχω δει στην συνέλευση σε εκπροσώπησης Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΚΕ. Εσείς ποτέ δεν το έχετε κάνει, ποτέ δεν έχετε παρευρεθεί. Λάβετε υπόψη τα δικαιώματα των ε, ανθρώπων και των μισθωτών και των δημοσίων υπαλλήλων θες, σας τα θέτω υπόψη και λάβετε υπόψη πολύ περισσότερο από το ιδιωτικό σας συμφέρον, το προσωπικό σας συμφέρον. Ο κύριος Θέρκας έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Βρισκόμαστε όπως είπε η κυρία Υπουργός, όχι μόνο μπροστά σε μια μεγάλη τραγωδία που συνέβη στην βιομηχανία Ταστρεϊν, αλλά μπροστά σε μια σημαντική προειδοποίηση. Προειδοποίηση που πρέπει να είναι για απόψε σημαντική υπόθεση, να μα κάνει να σκεφτούμε για το σύνολο των συντελεστών που συναπαρτίζουν μια κατάσταση απαράδεκτη συνολικά για την ανθρωπότητα και για τη δικαιοσύνη. Υπάρχουν εκατομμύρια εργαζομένων παγκόσμια που ασκούν τα καθήκοντά τους υπό όρους δουλείας χωρίς ε, οποιαδήποτε προϋπόθεση για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειάς τους. Θέλω να το κάνω και να το πω αυτό, διότι είναι σημαντική στιγμή αυτή για αυτά τα θέματα, χωρίς να ξεχνάμε και τα άλλα θέματα και τα άλλα ζητήματα. Είναι πολύ σημαντικό να υπενθυμίσουμε απόψε την ανάγκη να υλοποιηθεί η νομοθεσία του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, κυρίως οι οκτώ συμβάσει που είναι οι πιο σημαντικές και την ανάγκη να επεκταθούν αυτά παγκόσμια με νομοθεσία που θα διασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια. Όποια και να είναι η χώρα και θα προσέθετα όποια και να είναι και επιχείρηση. Αληθεύει ότι έχει πολλά όπλα και εργαλεία για να επεκτείνει αυτέ τι ανησυχίε, αυτά τα μελήματα για αυτέ τι συμβάσει του Διεθνού Γραφείου Εργασία. Δεν πρέπει μόνο να δίνουμε μαθήματα όμω, πρέπει να είμαστε υποδειγματικοί και να δίνουμε το καλό παράδειγμα. Υπάρχουν πολλέ ε, φωνέ που λένε ότι πρέπει να υποβαθμίσουμε και να ε, πάμε πιο κάτω στι προδιαγραφέ ε, για την υγεία και την ασφάλεια σε σχέση με του εργαζόμενου και ιδιαίτερα σε σχέση με τι μικρέ επιχειρήσει και πιστεύω ότι πρέπει να μας κάνουν να προβληματιστούμε όλα αυτά. Δεν είναι μόνο δουλειά μας, δεν μπορούμε να δίνουμε μαθήματα, πρέπει να δίνουμε το καλό παράδειγμα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος και τώρα για ένα λεπτό Γκόρενς παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, είμαστε συνυπεύθυνοι για αυτά τα οποία έλαβαν χώρα στο Μπαγκλαντές. Τα άτομα που δεν επιβίωσαν μετά την πυρκαγιά σε ένα τελειέ Παραγωγή σε ένα πράσινο τη ΔΑΚΑ είναι θύματα και ενό συστήματο που θα μπορούσαμε να το συνοψίσουμε με το γερμανικό σλόγγαν Γκάιτ στην Gai» ή «Τσιγκουνιά είναι μαγιά» ή επί το αρχαϊκότερον ακάλιστο ο άπλιστος». Υπάρχει μια φρενιτόδης αναζήτηση και του τελευταίου σέντ οικονόμηση για την αγορά ενό τη ΣΕΤ και αυτό παράγει, οδηγεί τους παραγωγούς ε, στι αναπτυξιόμενες χώρε να παράγουν όλο και πιο φθηνά και βέβαια επιβάλλουν κυρίω ε, στι γυναίκε που εργάζονται εκεί πάρα πολύ ε, απαράδεκτες ε, αμοιβέ δίνουν. Σίγουρα λείπουν ε, οι κανόνες που σέβονται τα κοινωνικά δικαιώματα, είναι ντροπή αυτό, αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε έτσι τα πράγματα και να βρούμε ελαφρυντικά. αν το fair trade και η θέληση να μπλοκάρουμε, να μποϊκοτάρουμε τις επιχειρήσεις που ε, δεν πληρούν αυτά τα ε, πρότυπα. Αν αυτό λοιπόν ε, μας βοηθήσει λίγο να, δεν μας βοηθήσει να βελτιώσουμε, θα μπορέσει παρόλα αυτά να θυμίσω ότι υπάρχουν εναλλακτικέ. Και έτσι θα αρχίσει να αντιστρέφεται και αυτή η λογική που, στην οποία οφείλεται και αυτή η καταστροφή που δεν είναι μεμονωμένη περίπτωση. De ευχαριστώ πρόεδρε. Ο πρέσβης ε, ε, του Μπαγκλαντές συζήτησε μαζί μας εχθές και επεσήμανε ένα γεγονός και ανέφερε και είπε ότι οι εργάτες της κλωστοϊφαντουργίας ε, εκείνοι που παράγουν αυτές τις φανέλες και τα ρούχα που εξάγονται στην Ευρώπη κάποιες δεκάρες μόνο εισπράττουν για την εργασία τους. Τα άτομα που εργάζονται στις ε, κλωστοϊφαντουργικές αυτές επιχειρήσεις είναι τα πραγματικά θύματα αυτής της κατάστασης. Ε, γίνεται, παράγονται αυτά τα ενδύματα, πολλούνται σε ε, υψηλές τιμές στην Ευρώπη και κάτι θα πρέπει να κάνουμε. Μπορούμε να έχουμε εθελοντικού χαρακτήρα συμφωνίες ή να υπάρχει και μια ετικέτα για αυτά τα προϊόντα. Όμως το Κοινοβούλιο απαιτεί όχι εθελοντικού χαρακτήρα, αλλά δεσμευτικού χαρακτήρα κώδικες για αυτές τις επιχειρήσεις. Θέλουμε υποχρεωτικού δεσμευτικού χαρακτήρα διατάξεις, ώστε να μπορούν με αυτές τις δεσμευτικές προϋποθέσεις και όρους να παράγουν αυτά τα ενδύματα. Πώς εκτιμάτε εσείς λοιπόν ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή την πρόταση. Πρόεδρε, πρέπει να λάβουμε υπόψη κυρίως ότι το Μπαγκλαντές είναι μια σταθερή δημοκρατία που καταβάλει πραγματικές προσπάθειες για να υλοποιήσει τις υποχρεώσεις της έναντι των δικαιωμάτων του ανθρώπου και εξαρτάται από το εμπόριο σε σχέση με τα κλαστοϊφοντεργικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να διατηρηθεί αυτή η πορεία. Αυτό το οποίο συνέβη με αυτή την πυρκαγιά ήταν πραγματικά δραματικό, μια τραγωδία. Δόθηκαν όμως διασφαλίσεις ότι θα υπάρξει σε βάθος εξέταση από τις αρχές του Μπαγκλαντές και υποστήριξη των οικογενειών των θυμάτων. Περισσότερα θα έπρεπε να γίνονται βέβαια όσο αφορά την κοινωνική περίθαλψη και τις κοινωνικές υπηρεσίες. Όμως υπάρχει βαθιά φτώχεια που πλήττει τη χώρα αυτή, το Μπαγκλαντές. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παράσχουμε κάθε βοήθεια στις αρχές ε, του Μπαγκλαντές σε αυτά τα προγράμματα ελέγχων ώστε να μπορέσει αυτή, να γίνονται αυτοί οι έλεγχοι αποτελεσματικά. Και έτσι με θελοντικές συνεισφορές ε, να μπορέσουν να αποζημιωθούν ε, οι οικοί των θυμάτων μέτρων. Όμως απορρίπτουμε τον υποχρεωτικό χαρακτήρα τέτοιου είδους ε, μέτρων. Επεκτείνουμε τα συλληπιτήριά μας στους συγγενείς και πρέπει να γίνει κάθε προσπάθεια να αποφευθούν τέτοιου είδους τραγωδίες στο μέλλον. Ευχαριστώ. Thank you. now one minute for Mr. Mr. Salvini. Κύριε Σαλβίνη, τελευταίος, ε, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μιλάμε για 112 νεκρούς και 100 ε, τραυματίες. Πρόκειται για κροκοδίλια δάκρυα και φταίμε εμείς οι Ευρωπαίοι γραφειοκράτες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δεν κάνουν τίποτα ε, για τις συνθήκες εργασίας αυτών των εργαζομένων που εργάζονται ε, για τις ε, μεγάλες πολυεθνικές με αμοιβή ένα δολάριο την ημέρα. Η Επιτροπή δεν θέλει στην ουσία να αλλάξει τίποτα. Δεν την ενδιαφέρει η σήμανση Made in. Ξέρετε τι κερδίζουν οι πολυεθνικές τους φορολογικούς παραδείσους. Χάνουν ε, πολύ εργαζόμενοι στην Λομβαρδία, στην Ιταλία, στην Ευρώπη, αλλά όλα τελειώνουν εκεί με την υποκρισία της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί για να κερδίσουμε μερικά δολάρια δεν μας ενδιαφέρει να χτίσουμε την Ευρώπη αλλά χτίσουμε την Ασία. Ο κύριος Κάσπαρη για τρία λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Εν μέρη βλέποντας τις τιμές αυτών των ενδυμάτων στην Ευρώπη για παράδειγμα, όπου για 3-4 ευρώ μπορεί να πάρει αγορά κανείς παντελόνια, jeans. Και όταν σκέφτομαι πώς πολλοί από τους συμπολίτες μας είναι ευγνώμονες ότι είναι δυνατόν δεδομένης της ε, ανεργίας και των χαμηλών μισθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορούν να αγοράσουν καν τέτοιου είδους παντελόνια, jeans. Ε, τότε σκέφτομαι ότι είναι λαϊκισμός ε, να υβρίζουμε τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αλλά πρέπει να ανταποκρινόμαστε στην πραγματικότητα ότι τα άτομα στην Ευρώπη, οι πολίτες στην Ευρώπη εποφελούνται από αυτή την παγκοσμιοποίηση. Παρ' όλα αυτά όμως πρέπει να συνεισφέρει η πολιτική για το εμπόριο να βελτιωθούν ε, οι διατάξεις και προδιαγραφές. Και το κάνουμε αυτό και με δεσμευτικές διατάξεις τη συμφωνία και το εμπόριο να συνεισφέρει έτσι ώστε αυτές οι χώρες όπου αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν δυσχερέστατη κατάσταση οι εργαζόμενοι σιγά σιγά να αναβαθμιστούν οι όροι απασχόλησής τους και αυτό θα είναι ένα μήνυμα της ανάπτυξης η κλωστοϊφαντουργία θα πρέπει να μετεξελιχθεί ε, όχι μόνο να μετεγκαθίσταται από τη μια χώρα στην άλλη μια και βλέπουμε ότι είναι μία από τις ε, βιομηχανίες που βρίσκονται στην αρχή μιας οικονομικής ανάπτυξης για κάθε χώρα και πρέπει να δούμε και τις θετικές πτυχές ε, για τους πολίτες ε, που συνεπάγεται μια τέτοια δραστηριοποίηση. Όμως ερωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι έκανε και κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τα τελευταία χρόνια ώστε εκτός της ε, εμπορικής πολιτικής να μεριμνήσει να υπάρξουν βελτιώσεις. Στην εξωτερική πολιτική λοιπόν να δραστηριοποιηθεί και να υποστηρίξει. Τι έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα στο πλαίσιο του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας επιτέλους όχι μόνο στο Διεθνή Οργανισμό Εμπορίου, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, στον ΠΟΕ, αλλά και αλλού να είναι δεσμευτικέ αυτές οι διατάξεις και προδιαγραφές. Τι έκανε πέρσι τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Διεθνέ Διεθνές Γραφείο Εργασίας επιτέλους να υπάρξουν δεσμευτικά μέτρα για την επιδιαιτησία και την επίλυση προβλημάτων. Γιατί πάντα υβρίζουμε την εμπορική πολιτική και γιατί δεν επομίζονται άλλοι τομείς ε, τις ευθύνε τους. Ε, ερωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποια μέτρα μέτρα έλαβε όσον αφορά τους φορείς για τις διεθνείς προδιαγραφές και διατάξεις ώστε να υπάρξουν καλύτερες προδιαγραφές για την εργασία και παραγωγή. Θα ήμουν ευγνώμων αν στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούσε να απαντήσει αυτά τα ερωτήματά μου. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε, σε διάλογο μεταξύ των επιχειρήσεων και των παραγωγών χωρών για τις ελάχιστες αυτές ε, προδιαγραφές. Όχι μόνο με την ε, κρατική επιβολή αλλά και εθελοντικά όπως ε, προβαίνουν αυτές οι χώρες. Το θέμα της εταιρική κοινωνικής ευθύνης αναφέρθηκε πολύ σχηδός. Ένας αποτελεσματικός διάλογος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρέπει να διεξαχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτέ τι χώρες για μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν οργανωτικά, για αποτελεσματικά συστήματα ελέγχου. Και άλλε χώρε θα μπορούσαν πολλά να μάθουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώ μπορούν να ελεγχθούν οι προδιαγραφέ αυτέ, αν τηρούνται και είναι σεβαστέ ή όχι. Θα ήμουν ευγνώμων αν μπορούσε να απαντήσει στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τι έχει γίνει για το ένα ή άλλο θέμα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριο για 1,5 λεπτό τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ως βουλευτής ε, και ως ε, εισηγητής συμμερίζομαι την οδύνη των ε, συγγενών των θυμάτων αυτών οι οποίοι πέθαναν με άσχημο τρόπο. 112 άτομα μεταξύ των 700 θυμάτων στο Μπαγκλαντές μόνο τελευταία δεκαετία και πραγματικά συμπάσχω. Ξέρω ότι το 50% της χώρας αυτής βασίζει σε εξαγωγές ειδών ένδυσης και σίγουρα και η κυβέρνηση έχει <clears throat> τη μισή ευθύνη, την άλλη την έχουν επιχειρήσει. Θα πρέπει λοιπόν αυτή την συζήτηση να καταγγείλουμε εταιρείε όπως είναι και η Walmart και η CNH ε, και η CNA και η H&M ε, που δεν έχουν αναβαθμίσει τις συνθήκες αυτά τα εργοστάσια. Ε, φεύγουν από το ε, Εδιμβούργο, φεύγουν από τη Γερμανία, οι επιχειρήσεις πηγαίνουν, δεν έχουν συναντήσει ούτε καν συνδικαλιστές που, που ζητούν εδώ και μήνες. Εγώ επίσης βλέπω ότι έχει γίνει κάποια πρόοδος με, τα, με τις διάφορες μάρκες, έχουμε κάποια πρωτοβουλία για ηθικό εμπόριο ή τη λεγόμενη πρωτοβουλία clean clothes, καθαρά ρούχα. Πάντως θα πρέπει να εφαρμοστούν στι πολυεθνικές και τα κριτήρια του ΩΣΑ, αλλά και τα κριτήρια σε ό,τι αφορά τι επιχειρήσει ε, και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όταν ο κύριο Μπαρνιέ προτείνει, και ελπίζω να το κάνει νωρίτερα, ε, την αναμενόμενη πρότασή του για την ε, διαφάνεια των εταιριών στην αλυσίδα εφοδιασμού και όταν συζητηθεί και ψηφιστεί δική μου πρόταση, θα πρέπει κανένα να πει ότι η κοινωνική εταιρική ευθύνη είναι προαιρετική. ακούγοντα το τι μα λέει το Μπαγκλαντέ, ε, πρέπει να αποδεχθούμε την κοινή ευθύνη και έτσι μόνο να σταματήσει η κατόμβη των θυμάτων. Σας ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Ο κύριος Φίσας έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρία Υπουργέ. Καταρχάς θα ήθελα να εκφράσω και εγώ τα συλληπιτήριά μου προς τις οικογένειες των θυμάτων αλλά και των τραυματιών των τραγικών συμβάντων των εργοστασίων και βιοτεχνών δημάτων στον Μπαγκλαντέ και στο Πακιστάν. Τεράστια ατυχήματα, δυστυχήματα που θα πρέπει να μα κάνουν να σκεφτούμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στηρίξει τι αναπτυσσόμενε χώρε, ευνοώντα και ενισχύοντα τι εισαγωγέ από αυτέ, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει αυτέ οι χώρε να πληρούν τα ελάχιστα, τα κατώτατα πρότυπα ασφάλεια, να σέβονται τα δικαιώματα των εργαζομένων, ε, να μην χρησιμοποιούν ε, ε, την παιδική εργασία, να σέβονται τα περιβαλλοντικά πρότυπα και κανόνε, ώστε να μην χρειαστεί να θρυνήσουμε περισσότερα θύματα λόγω αντίστοιχων δυστυχημάτων. Θα ήθελα να πω ότι πρόκειται για ένα ε, κοινωνικό και περιβαλλοντικό dumping σε πολλέ αντισώμενε χώρε, αυτό που ε, βλέπουμε. Όχι μόνο σε ιδιένδυση, αλλά και σε πολλέ άλλε επιχειρήσει και εργοστάσια. Αυτές οι καταχρηστικές ε, πρακτικές που κινούνται στο ε, περιθώριο ε, της νομιμότητας υπονομεύουν τα δικαιώματα και την υγεία των εργαζομένων και βέβαια βλάπτουν και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στους ευρωπαίους εργαζομένους. Πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επαγρυπνεί ώστε η διεθνής νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργασιακά δικαιώματα, το περιβάλλον να πληρούνται στις ανθρώπινες χώρες. Θα πρέπει να λάβουμε ριζικά μέτρα και να θέσουμε ως προϋπόθεση για την εισαγωγή προϊόντων κατασκευάσεων στις χώρες αυτές το σεβασμό αυτών των κατωτάτων προτύπων για την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος. Είναι κανόνες αυτοί και πρότυπα που εμείς εφαρμόζουμε στα προϊόντα τα οποία παρασκευάζονται εντός των συνόρων μας. Καταλήγοντας, ε, θα πω ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να επαγρυπνήσουμε για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ε, ασφάλεια των εργαζομένων σε αναπτυσσόμενες χώρες ε, και να αποφύγουμε τέτοιες τραγωδίες και δεύτερον προστατεύσουμε και τα δικαιώματα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και των ευρωπαίων εργαζομένων από αθέμητο ανταγωνισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Για 1,5 τώρα λεπτό, λέει ο Πρόεδρο, το λόγο έχει ο κύριο Μορέιρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επιτροπή, αγαπητοί συνάδελφοι, καθώ η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κύριο πελάτη όσον αφορά κλωστοϊφαντουργικά προϊόντα από τον Μπαγκλαντέ, έχουμε ειδικού ιδιαίτερου λόγου να ανησυχούμε για τι χείριστε συνθήκε απασχόληση των εργαζομένων εκεί. Μια και είμαστε γενναιόδοροι σε σχέση με τις ε, εμπορικές ε, προτιμήσεις ε, σε σχέση με το Μπαγκλαντές. Έχουμε κάθε δικαίωμα να απαιτήσουμε τέτοιου είδους καταστροφές να μην συνεχιστούν πλέον και προφανώς θα πρέπει να ληφθούν τα σωστά μέτρα ως απάντηση από τις αρχές του Μπαγκλαντές. Δηλαδή η υποστήριξη των οικογενειών των θυμάτων, η διακρύβωση των αιτίων της πυρκαγιάς, της πυρκαγιάς και των όσων ε, συνέβησαν σε αυτές τις ε, επιχειρήσεις. Αλλά αυτά είναι ένα μέρος μόνο των όσων πρέπει να γίνουν. Πρέπει να πετήσουμε από την κυβέρνηση της Μπαγκλαντές ε, τέτοιου είδους περιπτώσεις να μην επαναληφθούν. Πρέπει να είναι σεβαστή η νομοθεσία. Η επιθεώρηση εργασίας και οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται σωστά, ώστε σε σχέση με τις ε, επιχειρήσεις όσοι είναι υπεύθυνοι παραβιάσεων να προσάγονται στα δικαστήρια και να τιμωρούνται. Όμως ε, η κατάσταση αυτή είναι κάτι που από κοινού συμμερίζονται και η εισαγωγή αυτών των προϊόντων στην Ευρώπη που εκμεταλλεύονται τους χαμηλούς μισθούς ε, και εκμεταλλεύονται τους πιο φτωχούς που εργάζονται υπό τις πιο απαράδεκτες συνθήκες και εισάγουν αυτά τα προϊόντα αυτές οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Θα έπρεπε να απαιτηθούν εργασιακές συνθήκες που θα είναι ελάχιστο, ελάχιστο επίπεδο αποδεκτές ε, έστω. Θα πρέπει να είναι σεβαστές οι αρχές και οι υποχρεώσεις και η κοινωνική ευθύνη, εταιρική κοινωνική ευθύνη δεν λειτουργήσουν αυτά ως ήπια νομοθεσία, soft law, πρέπει να περάσουμε σε μέτρα σκληρής νομοθεσίας, hard law, με κυρώσεις και πρόστιμα, για να βελτιωθεί η ζωή των εργαζομένων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δύο λεπτά στη συνέχεια, κυρία Στρίφλερ. Donc, η τραγωδία που έγινε στα εργοστάσια ε, στο Πακιστάν και στο δείχνει πόσο αξιοθρύνεται είναι οι ασφαλεία. Στο Παγκλαντέ ε, συγκεκριμένα είναι ο δεύτερο εξαγωγέα ε, ειδών ένδυση μετά την Κίνα στον κόσμο. Λόγω των άθλιων ελληνών μισθών και ιδίω και λόγω τη παιδική και κοινωνική εργασία. Υπάρχει λοιπόν πάρα πολύ μεγάλη εκμετάλλευση. Μεγάλε πάντω δυτικέ αλυσίδε του Πρέτα Πορτέ πηγαίνουν εκεί για να παρασκευάσουν τα δήματά του. Λόγω λοιπόν τη αυτής ε, ε, της διεθνούς ε, της κοπτικής ραπτικής οδήγησε σε αυτή την τραγωδία στο Μπαγκλαντές. Όλοι βέβαια είναι υπεύθυνοι, οι εργοδότες που είναι συνηθισμένοι, αλλά οι Ασιατές επίσης που οι ασιατικές αρχές που είναι διεφθαρμένες. Αλλά πρέπει να θέσουμε όλους ενώπιον των ευθυνών τους και θα πρέπει να μην επιτρέψουμε να μειώνονται οι συνθήκες ασφάλειας και οι μισθοί. Ε, θα πρέπει να επιβληθούν κανόνες ασφάλειας στα εργοστάσια άμεσα και τα, μάλλον, ε, τα θύματα τέτοιων παραβάσεων, ε, τα θύματα από το μη σεβασμό από τις πολυαθλικές, θα πρέπει να αποζημιώνονται και θα μπορούν μάλιστα να προσφέρουν στη δικαιοσύνη της χώρας όπου ε, συνέβη η παράβαση. Θα πρέπει να υπάρχουν διεθνείς ε, φορείς ώστε να μπορούν να επιβάλλονται κυρώσεις σε επιχειρήσεις που παραβιάζουν την νομοθεσία. Και για να τα απαντήσουμε για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα πρέπει να πω ότι οι ίδιες οι πολυεθνικές είναι αυτές οι οποίες ε, οδηγούν στην εξόντωση ουσιαστικά της μικρομεσαίας επιχειρήσεις. Thank um, Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει για 1,5 λεπτό η κυρία Στάινμπρουκ. Μάλιστα. Επανειλημμένα σημειώνονται τέτοιου είδου καταστροφέ. Και όταν έχουν συμβεί, όλοι συγκλονίζονται και περνάμε μετά πάλι στην κανονική ημερήσια διάταξη μέχρι την επόμενη καταστροφή. Γιατί επειδή κάποιε επιχειρήσει δεν μπορούν να έχουν αρκετά κέρδη ή θέλουν ακόμα περισσότερο να συμπιέσουν του μισθού. Και έτσι εξοικονομούν κονδύλια από την προστασία την κοινωνική και την προστασία τη υγεία τίθεται το ερώτημα ποιοι είναι υπεύθυνοι για αυτές τις καταστροφές ε, και για αυτά τα ατυχήματα. Σαφώς οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων, οι ιδιοκτήτες αλλά και οι επιχειρήσεις εδώ στην Ευρώπη και εμείς ως πολιτικά υπεύθυνοι. Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να μπορούν να συμπιέζουν τις τιμές αλλά πρέπει να ελέγχεται από ποιου ε, προμηθεύονται τα εμπορεύματα αυτά και υπό ποιου όρου παράγονται αυτά. Κανείς δεν μπορεί να βρει προσχηματικά κάποιες δικαιολογίε ε, και όταν είναι έτσι θολό το πεδίο, εικόνα. Γι' αυτό πολλά πρέπει να γίνουν. Πρέπει ανεξάρτητα συνδικάτα επιτόπου να ενισχυθούν από εμά. Πρέπει να υπάρχει σωστή εφαρμογή των συμβάσεων του διεθνού Γραφείου Εργασίας. Καθαρές αλυσίδε εμπορευμάτων και βελτίωση των όρων απασχόλησης των εργαζομένων με ανεξάρτητες επιθεωρήσεις εργασίας και ελέγχου. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να τονίσει και να ενδυναμώσει την αρχή τη εταιρική κοινωνική ευθύνη. Απογοητεύομαι για το ότι η συντηρητική φιλελεύθερη πλειοψηφία δεν θέλει να υποστηρίξει την τροπολογία μας στην Ολομέλεια ώστε να υπάρχει σωστή προστασία και μ, περίθαλψη των θυμάτων. Μέχρι αύριο στο ξανασκεφτείτε μήπως αλλάξετε γνώμη. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Δύο λεπτά η κυρία Σνίμπε Πρόεδρε, θα ήθελα να συλληπιθώ τους ε, συγγενείς τους ε, οικείους των θυμάτων στα εργοστάσια του Μπαγκλατές. Θερμά συλληπιτήρια, πραγματικά είναι τεράστια τραγωδία να χάνει κανείς αγαπημένους του ανθρώπους με τέτοιου είδους συμφάντα πόσο μάλλον που αυτά τα περιστατικά ήταν προβλέψιμα. Γι' αυτό στηρίζω απολύτω το παρόν ψήφισμα, αλλά ταυτόχρονα θα, θα ήθελα να σε ψήσω την προσοχή στο γεγονό ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στι χώρε μέλη θα πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα, ούτω ώστε να αποφύγουμε μελλοντικά τέτοιε τραγωδίε. Και δεν νομίζω ότι αρκεί να εγκρίνουμε ψηφίσματα ή να διοργανώνουμε σεμινάρια ή να υπογράφουμε καταλόγου καταλόγους συλληπιτηρίων. Αλλά νομίζω ότι λόγω ακριβώς αυτού του τραγικού δυστυχήματος, λόγω της απώλειας τόσο πολλών ανθρώπινων ζώων, λόγω της παιδικής εργασίας, λόγω των ελληπών ελέγχων, και λόγω των κινδύνων που προκάλεσαν αυτό το ατύχημα νομίζω θα πρέπει να αντιδράσουμε ταχύτερα και θα πρέπει να διαρωτηθούμε τι είδου εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβάλλουμε, πώς συμβιβάζεται αυτό με το αίτημά μας ε, σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η υποχρέωση κοινωνικών ε, συνθήκων εργασίας δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε μεγαλόσχημα λόγια, αλλά να γίνει να εφαρμοστεί και στι στοχές χώρε. και εμεί ω σημαντικέ εισαγωγικέ χώρε θα πρέπει να συμβάλλουμε εδώ θετικά. Και αυτό δεν είναι μόνο υπό το πνεύμα τη παροχή βοήθεια προ τι χώρε αυτέ, προέλευση των εργαζομένων, αλλά είναι και ει όφελο των επιχειρηματιών ε, οι οποίοι ασφαλώ θέλουν να αποφύγουν τέτοιου είδου τραγωδίε και στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα 1,5 λεπτό για την κυρία Ρέγνερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμε κύριε Μπαρνιέ, αξιότιμοι εκπρόσωποι του Συμβουλίου. Όταν συζητούμε για τις φοβερές τραγωδίες στο Πακιστάν και στο Μπαγκλατές, δεν μιλούμε μόνο πραγματικά για αδιανόητα πλήγματα της μοίρα, αλλά πραγματικά για τρομακτική αμέλεια και πραγματικά αυτή είναι η άλλη όψη μιας πολιτικής του ανοίγματο της αγοράς. Όσο μακρύτερα βρίσκονται οι επιχειρήσεις, τόσο περισσότερο κινδυνεύουν οι εργαζόμενοι, ενώ η εργοδοσία παραβιάζει κατάφορα τα δικαιώματα των εργαζομένων. Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να, κρύβουν ε, πίσω από, κρύβονται πίσω από τις αλυσίδες της υπεργολαβίας. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια κοινωνική λογοδοσία εκ μέρους των επιχειρηματών ε, ε, για, όσο για εκείνου που αμφιβάλλουν για τη χρησιμότητα του ψηφίσματο, θα ήθελα να του παρακαλέσω να το σκεφτούν αυτό καλύτερα. Γιατί το ψήφισμα αυτό περιλαμβάνει κάποιε πολύ πρακτικέ και εφαρμόσιμε συμβουλέ. Δηλαδή, ότι οι πρεσβείες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα στο Μπαγκλαντές, θα πρέπει να ε, θα πρέπει να είναι ανοιχτέ για την κατάθεση προσφυγών ε, για τέτοιου είδους ε, ατυχήματα και ε, πραγματικά πρόκειται για μέτρα τα οποία έχουν ε, εγκριθεί από το Παγκόσμιο Γραφείο Εργασίας κλπ. Και άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρχουν άμεσα συνομιλητές στις ίδιες τις χώρες, ώστε να μην σχηματίζεται η εντύπωση ότι υπεκφεύγουμε τις ευθύνες όταν πρόκειται για χώρες οι οποίες είναι εξαιρετικά απομακρυσμένες από εμά. Ευχαριστώ πολύ και τώρα δύο λεπτά για την κυρία Σάιφη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Επίτροπε Μπαρνιέ, αγαπητοί συνάδελφοι. όπω και άλλοι συνάδελφοι, έτσι και εγώ θα ήθελα καταρχά να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου για τι οικογένειε των θυμάτων. Έχουν περάσει έξι χρόνια από το τελευταίο ατύχημα που είχαμε και 600 άτομα έχουν χάσει τη ζωή του σε πυρκαγιές, σε εργοστάσια εφαντουργία στο Μπαγκλαντέ. Στα 5.000 τέτοια εργοστάσια της χώρα, τελικά οι συνθήκε όλο και επιδεινώνονται. Πρέπει λοιπόν να εργαστούν οι ιδιοκτήτε των, των εργοστασίων αυτών μαζί με μηχανικού προκειμένου να καταφέρουν να εξασφαλίσουν την ασφάλεια και θα πρέπει πραγματικά να ε, καταδιώξουν του ε, ανεύθυνου ιδιοκτήτε των εργοστασίων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε το σημαντικότατο αυτό πρόβλημα και να επιφέρουμε μια λύση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί και πρέπει να βοηθήσει τον Παγκλαντές. Κύριε Πίτροπε, θα ήθελα να μιλήσω όμω και τη συμπεριφορά ορισμένων πολυεθνικών όπως το έπραξαν άλλωστε και άλλοι συνάδελφοι. Χωρίς να θέλω να μιλήσω με τρόπο λαϊκίστικο και να φέρουμε εδώ πέρα στον συνάδελφο Γκάσπερη, θα ήθελα απλώς να αναφερθώ στις εταιρείες Walmart, C&A, Gap, που έχουν συμμετάσχει σε συμφωνίες για την ασφάλεια των εργαζομένων, αλλά τελικά η ευθύνη βαρύνει τις εταιρείες αυτές. Το λέω πάρα πολύ συχνά. Στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μπορούν να διαδραματίσουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο προκειμένου να διαχειθούν καλύτερα οι σωστές συνθήκες εργασίας παγκοσμίω. Δεν μπορούμε να περιοριζόμαστε απλώς στο να καταγγέλουμε τον έναν τον άλλον, να καταδικάζουμε κάποιες συμπεριφορές. Θα πρέπει και εμείς να προωθήσουμε κάποιες λύσεις οι οποίες υπάρχουν και λειτουργούν στην πράξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Για 1,5 λεπτό κυρία Άντρες Μπαρέα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η περίπτωση του Παγκλατές μα δημιουργεί πολλέ ανησυχίες και θλίψη για, τα, για τους εργαζόμενους που έχασαν τη ζωή του και για την παραβίαση των δικαιωμάτων τους. Ε, ορισμένοι, 700 ε, εργαζόμενοι έχουν ε, πεθάνει τα τελευταία χρόνια τα συνδικάτα του Μπαγκλατές έχουν καταγγείλει τις συνθήκες εργασίας, τις ε, διακρίσεις εις βάρος των εργαζομένων. Οι Μπαγκλαντές είναι ο δεύτερος εξαγωγέας στον κόσμο στα, στην κλωστοϊφαντουργία, γιατί πάρα πολλές σημαντικές ε, μάρκες παράγουν στο Μπαγκλαντές που είναι πολύ πιο φτηνό. Αυτοί οι πολυεθνικοί θα πρέπει να γνωρίζουν την αλυσίδα της παραγωγής και οι διεθνείς συμβάσεις ε, υποχρεώνουν το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εκπληρώνουν τις, ε, τους κανόνες του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Επίσης υπάρχει μια εταιρική ευθύνη ε, και στην περίπτωση των ατυχημάτων τα, οι εργαζόμενοι θα έχουν το δικαίωμα να μπορούν να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη. Ευχαριστούμε πολύ και τώρα δύο λεπτά για την κυρία Αγγελίλη. Presidente. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριε Επίτροπε. Το ατύχημα στο εργοστάσιο της Ντάκα είναι απαράδεκτο. 112 νεκροί στις φλόγες και 200 τραυματίες, γυναίκες και νέοι άνθρωποι. Δεν είναι το πρώτο σοβαρό ατύχημα, αλλά είναι και άλλα τα οποία συνέβησαν μετά από λίγες ώρες αλλού. Το πρόβλημα λοιπόν είναι σοβαρότατο είναι σοβαρότατη η έλλειψη μετρών ασφαλείας, πανικός έλλειψη εξόδων κινδύνου, κλειστές έξοδοι, ελάχιστα μέτρα προστασίας από την πυρκαγιά. Στο Μπαγκλαντές ε, η ένδυση αντιπροσωπεύει το 80% των εξαγωγών, κυρίως προς τις Ηνωμένε Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λοιπόν σημαντικό σημείο τη Συμφωνίας Συνεργασίας ανάμεσα στην Μπαγκλαντές και στην Ένωση θα πρέπει να είναι τα δικαιώματα των εργαζομένων. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητήσει σεβασμό των επιπέδων διεθνών συμβάσεων για την προστασία της εργασίας από όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες παίρνουν μέρος σε διαγωνισμούς ή με υπεργολαβίες αναλαμβάνουν εξαγωγές από τον Παγκλαντέσου και να μην ξεχνάμε ότι η παραγωγή σε αυτή τη χώρα γίνεται για τις μεγάλες πολυεθνικές κυρίως. Θα πρέπει επίσης να γίνονται σεβαστές και οι εθνικές ρυθμίσεις για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων και θα πρέπει το Μπαγκλαντές για να συνεχίσει τις προσπάθειες για να μειώσει την εργασία των παιδιών, ένα φαινόμενο που υποβόσκει, κρυφίως θα έλεγα υπάρχει στη χώρα αυτή, αλλά δυστυχώς άνω το ενός εκατομμυρίου μικρών παιδιών ασκούν απασχολήσεις οι οποίες μάλιστα είναι και επικίνδυνες. Τελευταίος ο ο κύριος Μπέρμαν, αν δεν τον βλέπω στην αίθουσα όμως, οπότε περνάμε στην διαδικασία Cash ένας έχει ζητήσει το λόγο με τη διαδικασία Catch the Eye, ναι, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Μπαρνιέ, αγαπητοί συνάδελφοι, θα, πλέ, θα πρέπει η συζήτηση αυτή να είμαστε προσεκτικοί, ούτως ώστε να μην μπερδέψουμε τα αίτια ε, και τα αποτελέσματα. Γιατί από τη μία τα όσα συνέβησαν είναι πραγματικά τραγικά και εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας προς τους οικείους των θυμάτων. Αλλά ε, θα πρέπει να κάνουμε κάποιες διαφοροποίησεις γιατί έχουμε ξεκάθαρες αποδείξεις ότι εκείνες οι χώρες που είναι ενταγμένοι στην παγκόσμια οικονομία αναπτύσσονται καλύτερα οικονομικά από εκείνε που απομονώνονται. Και είναι γεγονό ότι οι κοινωνικέ ε, προδιαγραφέ ε, στι φτωχέ χώρε δεν είναι όπω ε, στη Δύση. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια ανοιχτή πρόσβαση για τα προϊόντα των χρόνων αυτών προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίω ότι δεν θα πρέπει να τηρούνται κοινωνικέ προδιαγραφέ. Αλλά αν διατυπώνεται το αίτημα να κλείσουμε τα σύνορα ή να προβαίνουμε σε υπερβολικέ ρυθμίσει, τότε θα πετύχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα. Ταυτόχρονα η Επιτροπή θα πρέπει να προσπαθήσει οι δικές μας επιχειρήσεις πραγματικά να επηρεάσουν τα πράγματα στον Παγκλαντές ούτε ώστε να τηρούνται κοινωνικές προδιαγραφές και ε, ε, οι, όσοι έχουν τα κονδύλια της αναπτυξιακής βοήθειας να βοηθήσουν τις χώρες αυτές όπως τον Παγκλατές να μπορούν να τηρούν τις ε, διεθνείς προδιαγραφές. Κύριε Τόρερ, ε, θέλετε να απαντήσετε, υπάρχει κάποιο ερώτημα προς εσάς. Το δέχεστε, μάλιστα. Κυρία Βάιλερ έχει το λόγο. Ε, κύριε Τόρερ, εγώ ήθελα να πάρω το λόγο λόγω της δικής σας παρέμβασης. Δεν καταλαβαίνω ότι κάποιος εδώ στο σώμα αυτό, ακριβώς λόγω της θετικής εμπειρίας που έχει κάνει η Ευρώπη με την εσωτερική αγορά, να θέλει να περιορίσει το διεθνές εμπόριο. Αλλά διεθνές εμπόριο, έτσι όπως το κανονούμε στην Ευρώπη, πάντοτε συνδέεται με την έννοια της ευθύνη όχι μόνο με την κοινωνική πολιτική και όχι μόνο με την αναπτυξιακή πολιτική, αλλά και με την ευθύνη των επιχειρηματιών ή των επιχειρήσεων που, ε, που έχουν την έδρα τους στην Ευρώπη και που μπορούν ε, να αγοράσουν σε χαμηλές ε, τιμές τα προϊόντα αυτά και που θα πρέπει να τηρούν τις διατάξεις της Σύμβασης ΑΕΛΟ. Και οι διατάξεις αυτές ακριβώς δεν τηρούνται. Γι' αυτό βεβαίως θα πρέπει να έχουμε ελεύθερο εμπόριο, αλλά με ένα πνεύμα ευθύνης. Ε, ε, κυρία συνάδελφε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δική σας παρέμβαση, γιατί μου δίνει τη δυνατότητα να πω ότι εγώ είμαι υπέρ του να τηρούνται αυτοί οι κανόνες αλλά δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεπάγονται επιπλέον ε, γραφειοκρατικά άχθη. Ε, και ε, εγώ κατάλαβα την εισηγήτρια ότι θέλει να θέσει ένα αμφιβόλο το μοντέλο της ελεύθερης αγοράς και θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και το δεύτερο σημείο είναι το εξής. Εγώ συμφωνώ ότι πρέπει οι εταιρείε να, είναι, να φέρουν κοινωνική ευθύνη. Αλλά ε, οι καταναλωτές ε, επίσης έχουν μια, ένα, τμήμα, ένα κομμάτι της ευθύνης. Ε, και ο κύριος Κασπάρη θέλει να σας απευθύνει ένα ερώτημα. Το δέχεστε. Ωραία λοιπόν. Αξιότιμα κύριε Τόιρερ ε, συμφωνείτε με μένα ότι μετά τη συζήτηση που μόλις είχατε με την κυρία Βάιλερ είναι προφανές ότι η, πολιτική εμπορία δεν μπορεί να επιλύσει από μόνη της το θέμα αλλά θα πρέπει να πιέσουμε ώστε όλοι οι τομείς της πολιτικής να συμβάλλουν θετικά ούτω ώστε επιτέλους να, να ρυθμιστούν θετικά τα ζητήματα ασφάλειας των εργαζομένων. Γι' αυτό δεν θα πρέπει πραγματικά να παραμείνουμε περιορισμένοι στον τομέα της πολιτικής εμπορίου, αλλά να συμπεριλάβουμε και τους άλλους τομείς. Απάντηση. Πράγματι, ε, εγώ θεωρώ ότι είναι ε, σεβαστή αυτή η ανησυχία ότι με τον τρόπο αυτό επιβαρύνεται υπερβολικά η πολιτική εμπορίου. Αλλά εμείς πάντοτε διατυπώσαμε το αίτημα να τηρείται η κυριαρχία, γίνεται σεβαστή η κυριαρχία και των τρίτων χωρών. Και αυτό ισχύει και για την περίπτωση του Παγκλαντές. Εμείς μπορούμε να υποστηρίξουμε βέβαια κάποιες πρόοδους στον Παγκλαντές υπό την έννοια της στήριξης των κοινωνικών προδιαγραφών. Θεωρώ ότι αυτό είναι ορθός δρόμος, αλλά πραγματικά αναμένουμε με το πώς ακριβώς θα απαντήσει η Επιτροπή όλα αυτά τα ερωτήματα. Ευχαριστούμε. Και τώρα θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Μπαρνιέ να μιλήσει εξ ονόματος της Επιτροπής. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας άκουσα πολύ προσεκτικά και εξ ονόματος της Κάθριν Άστον και της Κρυσταλίνα Ζωζίεβα που πήραν το λόγο πριν από λίγο θα ήθελα να δώσω και εγώ μια απάντηση αφού σας άκουσα πολύ προσεκτικά όλους. Καταρχάς, να επιβεβαιώσω και εγώ ότι και εμείς αισθανόμαστε ιδιαίτερη συγκίνηση και εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας για την πυρκαγιά αυτή, την τραγωδία αυτή που έπληξε το εργοστάσιο του στην Ασουλία του Μπαγκλαντές τον Νοέμβριο του 2012. 112 είναι τα άτομα που έχασαν τη ζωή τους, πολλοί νέοι, πολλές νέες γυναίκες. Δυστύχημα που όπως πολύ σωστά είπατε κυρίες και κύριοι βουλευτές στις παρεμβάσεις σας θέτει πολύ σωστά το ζήτημα των ε, κοινωνικών εργασιακών διατάξεων στα εργοστάσια της Νοτιοανατολικής ε, Ασίας. Σαφώς λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γίνανε διάφορες ε, έρευνες που καταλήγουν σε διαφορετικά συμπεράσματα, καμία όμως έρευνα δεν τίθεται κατά της γενικότερης διαπίστωσης ότι ε, είχαν παραβιαστεί σαφώς ε, οι διατάξεις ασφάλειας στο εργοστάσιο αυτό. Πριν από λίγο ένα συνάδελφος ακριβώς αυτό τόνισε ότι υπάρχει μία κοινή ευθύνη η οποία βαρύνει τελικά και τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Η ευθύνη λοιπόν αυτή βαρύνει και τους διευθυντές όμως του εργοστασίου αυτού στο Μπαγκλαντές το οποίο παραβίαζε τους βασικούς κανόνες όσον αφορά την ασφάλεια και όσον αφορά το εργασιακό δίκαιο και την κοινωνική του διάσταση. Όπως είπε και η Επίτροπος Ζορζίεβα πριν από λίγο, οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Τακάρ, η κυρία Λαμπέρτ για παράδειγμα το είπε ξεκάθαρα και την ευχαριστώ γι' αυτό, οι εκπρόσωποι τη Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν αντέδρασαν πάρα πολύ γρήγορα. Η υφιστάμενη συζήτηση καταδεικνύει ότι αναγνωρίζουμε όλο και περισσότερο το ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ασχοληθεί με το ζήτημα τη ασφάλεια στην εργασία όσον αφορά τα εργοστάσια των εμπορικών μας οικονομικών εταίρων και θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε αν θέλετε την ευκαιρία αυτή που έχουμε με την τραγωδία αυτή προκειμένου να καταφέρουμε επιτόπου να επιφέρουμε κάποιες πολύ σημαντικές βελτιώσεις. Στις 25 Ιουνίου του 2012 έχουμε πλέον ένα στρατηγικό πλαίσιο, ένα σχέδιο δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στο πλαίσιο αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να λαμβάνει δράση για να προωθήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα στην εξωτερική διάσταση της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής και ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμοστούν οι κατευθυντήριες γραμμές και αρχές των Εθνών όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στις επιχειρήσεις. Μετά από όλα αυτά τα οποία είπατε, ο κύριος Λάγκε, ο κύριος Κασπάρη και πολλοί άλλοι, ο Ρίτσαρτ Χάουιτ μεταξύ αυτών, η κυρία Βάιλερ, μετά τις παρεμβάσεις λοιπόν αυτές θα ήθελα να σας πω ότι και πολλές άλλες πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, εμπλέκονται στην ε, τραγωδία αυτή. Εγώ βρίσκομαι εδώ πέρα και συμμετέχω στη συζήτηση αυτή και αντικαθιστώ την κυρία Κρυσταλίνα Ζορζίεβα, αλλά και στα πλαίσια πραγματικά του χαρτοφυλακίου μου, αρμόδιος για την εσωτερική αγορά, δηλαδή για τις δημόσιες συμβάσεις, αλλά ασχολούμενος επίσης και με την εξωτερική διάσταση των οικονομικών μας σχέσεων, ασχολούμαι και με το ζήτημα της κοινωνικής ευθύνης των εταιριών, της λεγόμενης εταιρική κοινωνικής ευθύνης. Ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ως στόχο να προωθήσει τη νέα αυτή απέτηση, δηλαδή την εταιρική κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων. Το 2011 κάναμε μια σχετική ανακοίνωση και προτείναμε στο τέλος του 2012 ένα σχέδιο δράσης στα πλαίσια του ε, εταιρικού δικαίου, της διακυβέρνησης των επιχειρήσεων, της κοινωνικής ευθύνης και όλα αυτά βέβαια έχουν να κάνουν με τις δικές μας τις επιχειρήσεις ευρωπαϊκές, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός. Κυρία Βάλλερ θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να προωθηθεί μια πιο, ένα πιο ανθρώπινο, πιο ισότιμο εμπόριο και προσπαθούμε στα πλαίσια του πρώτου τριμήνου του 2013 να προωθήσουμε μια νομοθετική πράξη όσον αφορά την μη χρηματοπιστωτική διαφάνεια των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει δηλαδή να λογοδοτούν για τις δραστηριότητές τους όσον αφορά την κοινωνική ευθύνη, την κοινωνική ενσωμάτωση και το περιβάλλον. Στο ίδιο τώρα πνεύμα και κατά αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι δείχνω ότι δεν μιλάμε γενικά και αόριστα. Αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση επεξεργαζόμαστε ένα κείμενο το οποίο ήδη σας παρουσίασα όσον αφορά την διαφάνεια ανά χώρα ξεχωριστά προκειμένου οι 600 επιχειρήσεις μας είτε συμμετέχουν στο χρηματιστήριο είτε όχι, ασχολούνται πάντως με την εξόριξη, με την εκμετάλλευση του υπέδαφους και που ουσιαστικά έχουν πολλές σχέσεις με τις χώρες της Αφρικής και της Ασίας υπασχολούνται επίση με την εκμετάλλευση των δασών. Οι επιχειρήσει λοιπόν αυτέ οι ευρωπαϊκέ θα πρέπει να λαγοδοτούν τι ακριβώ κάνουν, ποιο πληρώνει τι και ποιον. Ζήτημα λοιπόν το οποίο θα συζητηθεί και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο των Υπουργών. Όσον αφορά τον Μπαγκλαντέ, η πρόοδηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων αποτελεί ένα από του ε, σημαντικού στόχου στρατηγική μα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει τη συνεργασία τη με την κυβέρνηση του Μπαγκλαντέ προκειμένου να ενταθούν οι πρωτοβουλίε αυτέ όσον αφορά το λιανικό εμπόριο, όσον αφορά την υφαντουργία και το τομέα τη ένδυση. Και το ίδιο είχε γίνει και με άλλε περιοχέ τη Νοτιοανατολική Ασία, όπου υπάρχουν κάποιε ανησυχίε. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε του υποστηρικτέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι οποίοι θέλουν περισσότερα κοινωνικά δικαιώματα και οι οποίοι επιτόπου διαδραματίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Σα επιβεβαιώνω επίση και το λέω ιδιαίτερα αυτό απευθυνόμενο στον κύριο Τόμα Μάνι, στον κύριο Μπέρντ Λάγκε, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει σύντομα μία έκθεση όσον αφορά τις πιο τραγικές, απαράδεκτες αν θέλετε, τις χειρότερες μορφές εμπορίου και εργασίες που πλήττουν πάρα πολλά παιδιά παντού στον κόσμο. Θα δημοσιεύσουμε την έκθεση αυτή τις ερχόμενες εβδομάδες. Όλοι συμφωνούμε, αν δεν κάνω λάθος, ως προς τα διδάγματα τα οποία μπορούμε να αντλήσουμε από την τραγωδία αυτή. Και γι' αυτό το λόγο λέω μία ακόμη φορά ότι η απάντηση που εμείς πρέπει να δώσουμε δεν μπορεί να είναι απλώς απλή, δεν μπορεί να προέλθει μόνο μέσα από ένα μέσο ή από μία εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειαζόμαστε την αποτελεσματική συνδυασμένη λειτουργία πάρα πολλών οργάνων. Χρειαζόμαστε μια οικονομική, πολιτική, πολιτισμική διπλωματία. Χρειαζόμαστε περισσότερο διάλογο. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα προγράμματα ανάπτυξης που θα πρέπει ουσιαστικά να προωθήσουν ακόμα περισσότερο την τήρηση συγκεκριμένων συνθήκων και όρων. Υπάρχει έπειτα και εμπορική πολιτική την οποία πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και πρέπει να προωθήσουμε ακόμα περισσότερο την κοινωνική ευθύνη, την εταιρική κοινωνική ευθύνη των δικών μας επιχειρήσεων. Συνεργαζόμαστε με πάρα πολλούς συναδέλφους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με τους ομολόγους μας στα κράτη-μέλη προκειμένου η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι πραγματικά συντονισμένη και αποτελεσματική. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να δώσω κάποιες πολύ σύντομες απαντήσεις στις παρεμβάσεις που γίνανε. Jean Lambert. Steinberg και οι δύο έχετε πάρα πολύ δίκιο όταν λέτε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξουν αποζημιώσεις προς τις οικογένειες των θυμάτων. Εμείς ελπίσουμε όπως το είπε και η κυρία Λάμπερτ, ότι η τριμερής διάσκεψη που έλαβε χώρα μεταξύ των, της εργοδοσίας των θρησκευτικών οργανώσεων θα καταλήξει τελικά σε μια απόφαση τηρώντας ε, το εργασιακό δίκαιο. Κάσπαρη, Στάινρουκ. Οι δύο αυτοί συνάδελφοι αναφέρθηκαν στον, στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, με την οποία έχουμε προφανώς μια σχέση προκειμένου να προωθήσουμε τους κανόνες ε, υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας. Στον Μπαγκλαντές, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας προωθούν προγράμματα για την επαγγελματική κατάρτιση και εμείς σε μια ανακοίνωση της, 15, της 15ης Ιανουαρίου του 2013 αναφερόμαστε στις ε, δραστηριότητες αυτές. Ο κύριος Κάσπαρη ενδιαφέρεται ιδιαίτερα πιστεύω για τα ζητήματα αυτά που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα. Σας υπόσχομαι λοιπόν ότι θα διαβιβάσω στην κυρία Άστον τις παρεμβάσεις σας καθώς επίσης και στον Επίτροπο Ντεγκούτε. Εξ ονόματός μπορώ ήδη να σας πω ότι συμφωνούν και θα συμφωνήσουν οι κύριες Κάσπαρη προκειμένου να ξεκινήσει μια συζήτηση με τις δικές σου υπηρεσίες και να προτεθούν τελικά κάποια βιώσιμα μέτρα και δράσεις. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εργασίας πραγματικά προωθεί μέτρα για την ασφάλεια της εργασίας. Υπάρχουν ε, πολλά εργοστάσια φαντουργίας στον Παγκλαντές, τα οποία δυστυχώς δεν έχουν ακόμα επικυρώσει τη σύμβαση αυτή. Θα διαβιβάσω πάντως τις ιδέες σας ε, στους συναδέλφους μου, καθώς επίσης και στους Επιτρόπους Άντορ και Ταγιάννη, των οποίων οι υπηρεσίες ε, εργάζονται, όπως και η δική μου υπηρεσία, για πολλές από τις πτυχές του ζητήματος που θίξατε εσείς. Αυτά είχα να σας πω εξ νόματος της κυρίας Κρυσταλίνα Ζιοζίβα, η οποία έπρεπε να αποχωρήσει νωρίτερα, επειδή έχει ανελημμένες υποχρεώσεις της Βρυξέλλης. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος του Συμβουλίου, η κυρία Κράιτον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη που πήραν μέρος στη συζήτηση. Νομίζω ότι η συζήτηση αυτή έδειξε ότι είμαστε όλοι αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να αποτρέψουμε μια επανάληψη των τραγικών συμβάντων του μηνός Νοεμβρίου. Ο κύριος Μπαρνιέ αναφέρθηκε στα περισσότερα από τα θέματα και με πολύ καλό τρόπο οπότε δεν θα ξαναπώ αυτά τα οποία μας είπε. Ξέρω ότι έχετε πολλή δουλειά μπροστά σας. Πάντως αρκετά μέλη έκαναν θετικά, θετικές προτάσεις και συστάσεις. Νομίζω λοιπόν ότι όλα τα μέλη θα πρέπει να σκεφτούν και επιπλέον προτάσεις για να μην επαναληφθούν, επαναλαμβάνω και εγώ, αυτά τα συμβάντα της Ντάκα και να μην χρησιμοποιηθούν βέβαια και σαν άλοθη για προστατευτικού τύπου μέτρα από πλευράς της Ευρωπαϊκής, από, από την Ευρωπαϊκή πλευρά. Νομίζω ότι με τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες και τις διμερείς συμφωνίες και μέσω του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας είμαστε σε θέση να βρούμε τρόπους έτσι ώστε να διασφαλίσουμε καλύτερα και υψηλότερα επίπεδα προστασίας για τους εργαζομένους στην χώρα αυτή. Αυτό το είπανε πολλά μέλη έχει σημασία από πλευρά Συμβουλίου να πούμε ότι εμείς θέλουμε μέσω του εμπορίου να δώσουμε κίνητρα προς τις χώρες αυτές έτσι ώστε να σεβαστούν τις βασικές απαιτήσεις και δικαιώματα αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος και τις ε, χρηστές αρχές διακυβέρνησης. Όπως είπα στις εισαγωγικές μου παρατηρήσεις ε, και μέσω του πλαισίου εμπορικών συμφωνιών έχουμε δυνατότητες στα πλαίσια αυτών των συμφωνιών να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τα οποία αναφέρθηκαν. Δεν θα επαναλάβω λοιπόν αυτά που είπε ο κύριος Μπαρνιέ. Νομίζω ότι ήδη θίξαμε σήμερα κάποιους τρόπους προώθησης μιας ισορροπίας ανάμεσα στο εμπόριο, το περιβάλλον και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Νομίζω ότι Όλοι θα πρέπει να συνεργαστούμε με τον ILO, με το Διεθνές ε, Γραφείο Εργασίας, Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, γιατί έτσι θα διασφαλίσουμε κατάλληλες συνθήκες απασχόλησης σε όλες τις χώρες με τις οποίες έχουμε εμπορικές σχέσεις. Ευχαριστώ πολύ. Κλείνει η συζήτηση αυτή. Υπάρχουν έξι προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο το 12η μεσημβρινή. Τώρα περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Η δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την κατάχρηση των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις επιπτώσεις της πολιτικές διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Θα ξεκινήσουμε με την δήλωση από πλευράς του Συμβουλίου. Την δήλωση θα κάνει η Υπουργός Κράιτον. Ευχαριστώ Πρόεδρε.